Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Σας εύχεται ο Πρόεδρος. Καλώς ήρθατε στην κοινή αυτή δημοσία ακρόαση με το ερώτημα μήπως ήρθε η ώρα να ξαναδούμε την θερινή ώρα. Πρόκειται για κοινή ακρόαση, όπως είπα, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας και μεταφορών και τουρισμού. Λόγω ασθενείας ή και άλλων ελληνικών υποχρεώσεων, οι δύο άλλοι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών επιτροπών δεν μπορούν να προσέλθουν. Θα ήθελα όμως να καλωσορίσω εγκαρδίως τους διακεκριμένους ομιλητές μας και θα ήθελα επίσης να απευθύνω το καλό, ορίσατε στον κύριο Πέτερ Σίλαρ, μέλος της τσεχικής γερουσίας και μέγα υπέρμαχο της κατάργησης θερινής ώρας. Έχει κάνει και μια εκστρατεία και ένα έγγραφο επομένως που ε, ε, επιγράφεται στα αγγλικά «For only one time» Καλώς ορίσατε λοιπόν. Πριν δώσω το λόγο τώρα στους διακεκριμένου ομιλητές να σας προσκαλέσω να τηρήσετε ενός λεπτού σιγή περί της μνήμης των θυμάτων της τραγωδίας, αεροπορικής τραγωδίας με την πτώση του γερμανικού αεροσκάφους πάνω από τι Γαλλικές Άλπεις. you Σας ευχαριστώ. Στο πρώτο μέρος της η ακρόαση θα ασχοληθεί με θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Να δώσω το λόγο πρώτα στην κυρία Χίλ Κασάδο, επικεφαλής του Τμήματος Διαθεσμικών Σχέσεων της Αρμόδιας Γενικής Διευθύνσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 10 λεπτά, κυρία μου. Thank you very much, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, κύριοι βουλευτές. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σας ευχαριστεί που μας ε, δίνετε τη δυνατότητα να ε, συμμετάσχουμε σε αυτήν την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να, κάνω ένα, να σας δώσω ένα πλαίσιο όσον αφορά αυτό το νομοθέτημα το οποίο ήδη το 2001 ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύο φορές το χρόνο αλλάζει το ρολόι σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το χειμώνα στο καλοκαίρι και από το καλοκαίρι, δηλαδή από τη θερινή ώρα, στην ε, χειμερινή ώρα. Η αρχή έγινε στη δεκαετία του 60 και στη δεκαετία του 70 στις περισσότερες ε, χώρες. Αλλά οι αλλαγές ε, δεν γινόντουσαν πάντα ταυτόχρονα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την δημιουργία της εσωτερικής αγοράς κατέστη σαφές ότι μια εναρμονισμένη προσέγγιση των ε, διαφορετικών ρυθμίσεων της τερινή ώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ε, έπρεπε οπωσδήποτε να υπάρξει η νομοθεσία σε ενωσιακό επίπεδο υπάρχει έτσι ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει καλά η εσωτερική αγορά δηλαδή να λειτουργήσει μέσω ε, σαφώς καθορισμένων ε, στιγμών αλλαγής δύο φορές το χρόνο. Η θερινή ώρα ε, είχε ήδη εισαχθεί από κράτη-μέλη σε εθνικό επίπεδο. Επομένως, η μόνη απόφαση η οποία ελήφθη σε ενωσιακό ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν να καθοριστεί η συγκεκριμένη ημερομηνία και η ακριβή στιγμή που αυτή η αλλαγή θα ελάμβανε χώρα. Η οδηγία ε, η οποία βρίσκεται εν είναι αυτή που όπως ανέφερα προηγουμένως ε, άρχισε να ισχύει το 2015 ε, και είχε μάλιστα ζητηθεί συγκεκριμένα από 15 χώρες μέλη. Ε, πρόκειτο για χώρες οι οποίες είχαν ήδη παρατηρήσει ότι υπήρξαν, υπήρχαν δυσκολίες στην εσωτερική αγορά ε, λόγω ακριβώς της διαφοροποιημένης εφαρμογής της θερινής χώρας από, μια, από τη μία χώρα στην άλλη. Ας πούμε οι, οι επικοινωνίες, οι μεταφορές είχαν αντιμετωπίσει προβλήματα και επομένως χρειαζόταν συντονισμός όσον αφορά το θέμα αυτό. Σύμφωνα με την την ε, οδηγία αυτή του 2001 η Κομισιόν υπέβαλε έκθεση ήδη το 2007 ε, όσον αφορά τον αντίκτυπο της ε, θέσης σε ισχύ αυτής της οδηγίας. Εκεί χρησιμοποιήθηκαν κάποιες πληροφορίες που είχαν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω μελετών αλλά και από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Τα περισσότερα κράτη-μέλη αυτό που έκαναν ήταν στην ουσία ε, να έρθουν σε επαφή και να διαβουλευθούν με διάφορους κλάδους, με τους γεωργούς, ε, με τις ε, μεταφορές, με την υγεία κτλ. Βάσει των ευρημάτων αυτών των διαβουλεύσεων, ας πούμε στην, στην αναφορά αυτή, ε, αναφέρεται ότι στον τομέα της ενέργειας ε, οπωσδήποτε υπήρχαν κάποιες ε, εξοικονομήσεις που ωστόσο όμως δεν ήταν πολύ μεγάλες. Όσον αφορά την οδική ασφάλεια, υπήρχαν κάποιες χώρες όπως η Εστονία ή η Πορτογαλία ας πούμε, που έκαναν κάποιες συγκεκριμένες έρευνες για τα θέματα αυτά. Συνεπέραναν δε ότι δεν υπήρχαν πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις λόγω της αλλαγής ε, και της εφαρμογής της θερινής ώρας. Στον τομέα της ε, υγείας παρατηρήθηκαν κάποιοι, ε, παρατηρήθηκε κάποιος αντίκτυπος αλλαγή του ε, βιορυθμού, ε, του ρυθμού του ύπνου, λόγω της αλλαγής της ώρας. Ωστόσο, δεν μπορούν οι αλλαγές αυτές να θεωρηθούν ιδιαίτερα σημαντικές. Επομένως, ε, στην μελέτη του 2007 το συμπέρασμα ήταν ότι η εφαρμογή της θερινής ε, ώρας ε, ήταν καλή έτσι ώστε να ενθαρρυνθούν οι δραστηριότητες αναψυχής το βράδυ και ότι υπήρχαν και κάποιες εξοικονομήσεις ενέργειας και ότι, εν πάση περιπτώσει, μικρά ήταν τα αρνητικά αποτελέσματα αποτελέσματα και ο αρνητικός αντίκτυπος της ε, θερινής ώρας. Πέρσι, το 2014, η Κομισιόν έκανε μια άλλη ε, μελέτη Παρήγγειλε λοιπόν μία μελέτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να δει ε, ε, τον ενδεχόμενο αντίκτυπο ε, επί της εσωτερικής αγοράς της μη εναρμονισμένης θερινής ώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα συμπεράσματα ήταν ότι εάν δεν είχε υπάρξει αυτή η εναρμόνιση θα είχαν υπάρξει οπωσδήποτε κάποια επιπλέον κόστη όσον αφορά την ενέργεια, όσον αφορά τις μεταφορές ή και το διοικητικό ε, κόστος. Ε, γενικά πάντως η μελέτη δεν περιέλαβε σενάρια ε, για περίπτωση ακύρωσης της ανέρεσης της τερινής ώρας. Therefore, on the basis of this... Λαμβάνουμε λοιπόν υπόψη μας αυτές τις ε, οδηγίες και τον τρόπο με τον οποίο ε, εφαρμόστηκε η οδηγία του 2001 και συμπεράναμε τα εξής. Εάν καταργούσαμε αυτήν την εναρμονισμένη θερινή ώρα, ε, τότε θα δημιουργούνται ε, ε, πολλά προβλήματα όχι μόνο στους πολίτες αλλά και στις επιχειρήσεις. Και επομένως θα τελειώσω αναφέροντας κάτι που είπα στην αρχή. Η οδηγία ε, είναι ακριβώς ένα εργαλείο εναρμονισμένης λειτουργίας και στόχο έχει την καλή εναρμονισμένη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Κάποια κράτη-μέλη ε, σήμερα έχουν... Ε, ε, συγγνώμη, μέχρι τώρα τα κράτη-μέλη επισήμως δεν έχουν ζητήσει κατάργηση της θερινής ώρας, επομένως θεωρούμε ότι η εφαρμογή αυτής της θερινής ώρας θεωρείται προσήκουσα. Να τελειώσω λέγοντας και υπενθυμίζοντας μάλλον ότι ακριβώς αυτό το Σαββατοκυριακό, την Κυριακή, θα προχωρήσουμε τα ρολόγια μας, θα βάλουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία μου. Να ακούσουμε άλλη μια παρέμβαση και μετά να ακούσουμε έναν αριθμό ερωτήσεων που δεν απευθύνονται στις δύο αυτές παρεμβάσεις. Να δώσω το λόγο λοιπόν σε άλλο προσκεκλημένο μας, τον κύριο Λότον, που είναι σύμβουλος ασφάλειας μεταφορών από το Ενωμένο Βασίλειο. Έχει το λόγο αγαπητή κυρία για 10 λεπτά. Thank you very much, Mr. Chairman. Oh, that's better. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, λέγομαι Brian Lawton, TRL, Transport Research Laboratory. Είμαστε ιδιωτικοί εταιρεία. Ιδιωτικοποιηθήκαμε το 1996. Δεν έχουμε, δεν κατανέμουμε μερίσματα, όποια κέρδη κάνουμε τα ε, επενδύουμε στην έρευνα. Παραμένουμε έτσι ανεξάρτητοι. Εμείς ε, βρισκόμαστε και πίσω από κάποια από τα τεστ αυτοκινήτων που βλέπετε μια φωτογραφία εκεί. Ας αρχίσουμε με τα βασικά λοιπόν. Βλέπετε ένα πίνακα στο χάρτη υπάρχουν οι διάφορες ε, ζώνες, βεβαίως ο ήλιος ανατέλει στα ανατολικά και ε, στη δύση. Άρα, όσο πιο ανατολικά είσαστε, τόσο πιο νωρίς εικόνεστε. Όπως εξήγησε η Βικτόρια πριν, θα γνωρίζετε βέβαια ότι την άνοιξη βάζουμε το ρολόι μία ώρα μπροστά και το αυθινόπορο μία ώρα πίσω. Spring forward, fall back. Έτσι τα λέω εγώ για να τα θυμούμε στα αγγλικά. Τώρα, δέστε εδώ, η Ισλανδία δεν αλλάζει από την ώρα Greenwich. Βλέπετε ότι είναι στην ίδια ε, ζώνη. Το ίδιο με την Βρετανία και την Πορτογαλία. Υπάρχουν ορισμένε αφρικανικέ χώρε, εκεί βλέπετε στο βάθο, στο κάτω μέρο δηλαδή, όπω την Ισία και η Αλγερία, που και αυτέ δεν αλλάζουν. Όμω οι περισσότερε ευρωπαϊκέ χώρε αλλάζουν. και αυτό το λέμε θερινή ώρα DST, Daylight Saving Time. Ο λόγος για τον οποίο αλλάζουμε την ώρα είναι για να εκμεταλλευτούμε καλύτερα το περισσότερο φως της ημέρας το καλοκαίρι και το αντίθετο το χειμώνα. Αυτός ο τίτλος Daylight Saving Time, δηλαδή ώρα εξοικονόμησης ηλιακού φωτό. Δεν μπορείτε να εξοικονομήσετε το ηλιακό φω, βέβαια δεν μπορείτε να το βάλετε σε ένα μπουκάλι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μα. Σήμερα έφυγα εγώ από το σπίτι μου όταν ήδη είχε φω. Όταν θα επιστρέψω στο σπίτι μου θα είναι ήδη σκοτεινά από ώρα. Αν μπορούσα να αλλάξω το ωράριο θα μπορούσα να ταξιδέψω και φεύγοντα και επιστρέφοντα με φω. Τώρα από την άποψη της ασφάλειας των μεταφορών, γιατί έχει σημασία αυτό υπάρχει λιγότερος κίνδυνος συγκρούσεων, ιδίως για ποδήλατα και πεζούς, όταν, είναι, όταν υπάρχει το φως της ημέρας και όχι βέβαια όταν είναι σκοτάδι. Έτσι λοιπόν τα σκοτεινά πρωινά είναι κακά για την τροχιά κυκλοφορία, αλλά τα φωτεινά βραδινά είναι καλύτερα. Υπάρχει λοιπόν κάτι το οποίο εξορροπεί το άλλο. Βέβαια υπάρχει και μεγαλύτερη δραστηριότητα στους δρόμους το απόγευμα και το βράδυ και το καθαρό αποτέλεσμα τελικά είναι ότι αλλάζοντας την ώρα έχουμε λιγότερες συγκρούσεις το βράδυ, περισσότερες το πρωί, αλλά όχι τόσο, τόσο περισσότερες το πρωί, ώστε να ανατρέπεται το θετικό αποτέλεσμα που έχουμε το βράδυ. Άρα εδώ υπάρχει ένα πλεονέκτημα. Για να εξηγήσω λίγο περισσότερο. Κάποια παλιά δεδομένα από τη Μεγάλη Βρετανία από το 2009 στην περίπτωση αυτή δεν το επέλεξα επίτηδες ε, το slide αυτό, αλλά για να στηρίξω κάποιο επιχείρημα, αλλά το βρήκα εύκολα. Βλέπετε τον αριθμό των απολειών, δηλαδή των ε, θανάσιμων ζώων, των θανάσιμων ε, δυστυχημάτων ανάμεσα σε... Βλέπετε τον πίνακα τέλο πάντων, βλέπετε δεξιά μέχρι τα 11 και 12 και και βλέπετε ότι 8 με 9 το πρωί υπάρχει μια κορύφωση και 3, 4, 5, 6 το βράδυ. Με την θερινή ώρα μειώνουμε την κορύφωση αυτή στο δεξί μέρος. Θα έχει μια αύξηση η κορυφή στο αριστερό πλευρό της ε, διαφάνειας, αλλά συνολικά θα υπάρχει μείωση. Υπάρχουν τώρα και μερικά άλλα στοιχεία. Το αποτέλεσμα είναι λίγο πολύ ομοιόμορφο σε όλη την ε, Ένωση. Όμως όσο πηγαίνετε προς βοράν είναι λιγότερες λιγότερα τα ωφέλη, διότι είναι διαφορετικό εκεί το καλοκαίρι και ο χειμώνας από ό,τι είναι στην υπόλοιπη. Στο νότο δεν έχετε επίσης μεγάλη διαφορά. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, ακόμα και το χειμώνα, έχετε 10 ώρες φως με την ημέρα. Μέσα τώρα στις ίδιες τις ε, ε, ώρες μέσα στις ίδιες ζώνες ώρων, αν είσαστε προς τα ανατολικά της ζώνης ώρας, έχετε μεγαλύτερη ωφέλεια από ό,τι αν είστε στα δυτικά. Γνωρίζω καλύτερα τα πράγματα βέβαια για τη Μεγάλη Βρετανία, για αυτήν θα μιλήσω τώρα και θα μιλήσω και ε, μετά για ορισμένες από τις εμπειρίες ε, της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Ε, Στην Βρετανία λέμε αντί να αλλάξουμε για μια ώρα το καλοκαίρι, γιατί να μην αλλάξουμε δύο ώρες, να μην βάλουμε το ρολόι δύο ώρες μπροστά και γιατί να μην βάλουμε τη θερινή ώρα ολόκληρο το χρόνο. Ανάμεσα στο 1968 και στο 1971 λοιπόν μείναμε στο GMT 1, δηλαδή αυτό που αντιστοιχεί στην υπηρετική νυχτερινή ώρα, στην ε, ε, ε, χειμερινή ώρα δηλαδή, Και μέσα στα περιθώρια αυτά είχαμε 12% λιγότερους θανάτους στο, ε, από ατυχήματα στον δρόμο. Αν μείνουμε δηλαδή σε standard time όλο το χρόνο μπορούμε να σώσουμε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές ή να γλιτώσουμε πολλούς τραυματισμούς. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί καμιά παρηγοριά για αυτούς οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους ή συγγενείς τους τις πρωινές ώρες. Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιον και να του πείτε όμως να, αν δεν είχαμε αλλάξει την ώρα, εσύ θα είχε σωθεί ή δεν θα είχε σωθεί αντιστοίχω. Δεν μπορεί κανεί να εντοπίσει ακριβώ τα θύματα. Βέβαια, τα πράγματα έχουν αλλάξει από το 1971. Πιο πρόσφατα, το 2009, εξετάσαμε ξανά το θέμα και εξετάσαμε ιδίω αυτό που λέμε single-double summertime, δηλαδή να πάμε GMT συν το χειμώνα και GMT συν 2 το καλοκαίρι. Αυτό μας λέει ότι υπολογίζουμε δηλαδή θα έχουμε 80 θανάτους λιγότερους το χρόνο και 120 βαριούς τραυματισμούς λιγότερους. Αν δούμε τη γεωγραφία της Μεγάλης Βρετανίας πάλι τα αποτελέσματα ποικίλουν. Στη Σκοτία που είναι στο βορρά δηλαδή τι ερώτημα αν θα υπάρχει καμιά ε, ωφέλεια. Και όσο πιο δυτικά πηγαίνει κανείς τότε θα υπάρχουν πάλι περισσότερα θύματα. Τώρα άλλε ευρωπαϊκέ ευρωπαϊκές Η Πορτογαλία άρχισε ε, να, εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Ώρα το 1966 και το 1992. 96 Έχουν όμω περισσότερε ώρε, είναι λοιπόν φω το πρωί και το βράδυ. Ο λόγο λοιπόν για τον οποίο έκαναν την αλλαγή δεν ήταν η οδική ασφάλεια. Στη Σουηδία τώρα υπήρχε κάποια υποψία ότι ο αριθμός των συγκρούσεων θα άλλαζε, θα ανέβαινε ή θα έπεφτε μετά από την αλλαγή της ώρας. Έγιναν όμως κάποιες μελέτες που τελικά δεν έδειξαν καμιά αλλαγή στον αριθμό των συγκρούσεων. Ούτως ή άλλως οι άνθρωποι ξυπνούσαν νωρίς με το φως του ήλιου. Στη Γερμανία από την άλλη μεριά όταν άρχισε να επιβάλλεται η θερινή ώρα θεώρησαν ότι θα μειωθεί ο αριθμός των ατυχημάτων Είδαν όμως ότι τελικά αυξήθηκε, διότι το έξτρα, οι έξτρα ώρες φως σήμαινε ότι οι άνθρωποι κυκλοφορούσαν περισσότερο και τελικά υπήρχαν περισσότερες συγκρούσεις και ατυχήματα. Η Βικτόρια μίλησε ήδη για μια πιο πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από αυτήν που βλέπετε στην οθόνη τώρα και που λέει ότι ο κόσμος δεν αντιδρά τόσο πολύ στην αλλαγή της ώρας κάθε καλοκαίρι. Η τελευταία, ε, το 1995 δηλαδή, προ 20 τη της ε, Γεωργικής Συμβουλευτικής Υπηρεσίας λέει ότι θα υπάρχουν έξτρα ωφέλη εάν η Βρετανία ακολουθήσει την κεντρική ευρωπαϊκή ώρα. Θεωρούν ότι θα είναι η καλύτερη επιλογή από την άποψη της οδικής ασφάλειας. Συνοψίζω λοιπόν. Μα αρέσουν τα φωτεινά πρωινά, είναι καλά για την οδική κυκλοφορία, μα προτιμούμε ακόμα περισσότερο τα φωτεινά βράδια. Υπάρχει ανησυχία ότι ίσως αν, ε, με, ε, με τη θερινή ώρα να αυξηθεί, να αυξηθεί η κυκλοφορία ούτως ή άλλως. υπάρχουν κάποιοι άγνωστοι και το περιβάλλον είναι πολιτικά κάπως φορτισμένο. Έτσι λοιπόν τήρησα και το όριο των 10 λεπτών. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση, για την παρουσίαση που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουμε τώρα χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων και απαντήσεων. Από τους δύο πρώτους, ε, δηλαδή απαντήσεις από τους δύο πρώτους ομιλητές. Ανοίγω λοιπόν τον κατάλογο και πρώτη ε, λαμβάνει το λόγο η κυρία Νίπλερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ πρώτα την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και τον εμπειρογνώμονα. Να μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση. Προέρχομαι από τη μεγαλύτερη χώρα μέλος, δύο φορές το χρόνο ο κόσμος αγανακτεί, διότι θεωρεί αυτή την ε, αλλαγή της ώρας μια επιβάρυνση και μας ζητούν ξανά και ξανά να αναλάβουμε κάποια πρωτοβουλία για να καταργηθεί αυτή η θερινή ώρα. Εγώ βέβαια γνωρίζω και απευθύνομαι τώρα στην εκπρόσωπο της Κομισιόν και έχετε δίκιο ότι δεν είναι ευρωπαϊκό θέμα. Εσείς μιλήσατε για την οδηγία και το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να συντονιστεί η θερινή ώρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι βέβαια κατά τα άλλα θέματα, θέμα μάλλον των χωρών μελών αν θα επιλέξουν τη θερινή ώρα ή όχι. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, πολλούς τους δυσαρεστεί. Αυτή η θερινή ώρα. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έπρεπε να κάνει και κάποια έρευνα ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις της κατάργησης της θερινής ώρας. Θα είχε μεγάλη σκοπιμότητα κάτι τέτοιο. Δεύτερη ερώτηση, η δεύτερη παρατήρηση συνδεδεμένη με ερώτηση για τον εμπειρογνώμονα, για τον τομέα των μεταφορών. Εσείς εξηγήσατε λεπτομερώς πως εξελίσσεται η κατάσταση σύμφωνα με τις δικές σας ε, εμπειρικές παρατηρήσεις. Ακούω ότι ιδίως η τροποποίηση των ορολογιών προγραμμάτων των τρένων κοστίζει, κοστίζει πολλά λεφτά, διότι δύο φορές το χρόνο αναγκάζονται να αλλάξουν τα δρομολόγια όλων των τρένων και αυτό προκαλεί σημαντικό κόστος. Υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία γι' αυτό. Επίσης, ποιες είναι οι επιπτώσεις που έχει η θερινή ώρα στον βιορυθμό. Πάλι την προηγούμενη εβδομάδα έλαβα επιστολές από γιατρούς που μου μιλούν για την επίπτωση της θερινής ώρας στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Πρόκειται για μια ατελείωτη επιβάρυνση εν τέλει. Αυτό ήθελα να πω. Θα θέσω μετά άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τους βιορυθμούς μετά, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Ρόιλ. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, επίσης, κύριε και κύριοι, χαίρομαι πολύ που κατέστη επιτέλους δυνατόν να διεξαχθεί ακρόαση για το θέμα αυτό. Αυτό σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά εγκύπτει στο θέμα αν είναι καλό ή κακό. Αν είναι καλή ή κακή αυτή η υπόθεση της τερινής ώρας. Η πρώτη φορά που είχα ασχοληθεί είναι πριν από πολλά χρόνια και μιλήσατε πριν για αυτή την ε, μελέτη του 2007. Να ε, μελετήστε την έκθεση αυτών που περιλαμβάνει, που περιλαμβάνει τις συμβολές πολλών χωρών μελών. Έχει πολύ χιούμορ αυτή η οδηγία, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια απόλυτη ανοσία, διότι ο καθένας γράφει ό,τι του έρθει στην ουσία μη θέλοντας να ασχοληθεί. Προσπαθήσαμε μετά να ρωτήσουμε και τις χώρες μέλη, οι οποίες επίσης δεν απάντησαν τουλάχιστον όχι με ακρίβεια. Και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε άλλη μελέτη πρόσφατα. Δεν ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε επιστημονικά κριτήρια. Εγώ πραγματικά αγανακτώ με την ιδέα ότι ξοδεύονται χρήματα για τέτοιου είδους μελέτες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μετά από την ακρόαση πρέπει να αναρωτηθούμε πώς θα αποκτήσουμε ασφαλή, αξιόπιστα δεδομένα. Δεν αρκεί ο κόσμος να λέει ότι θέλω κάτι να αλλάξει. Πρέπει να γνωρίζω και γιατί. Ακούω ένα επιχείρημα τώρα ότι στην ε, οδική κυκλοφορία θα υπάρξουν περισσότερα ατυχήματα και περισσότερη νεκροί. Αυτό είναι ένα επιχείρημα το βασικό επιχείρημα όλων είναι ότι θα πρέπει να γίνει πανευρωπαϊκά, με συντονισμό. Βεβαίως και πρόκειται ακριβώς γι' αυτό. Δεν έχει νόημα μια χώρα μέλος να πει ναι και η άλλη όχι. Έχω και μια διαδικαστική ερώτηση που θέλω να απαντηθεί. Ελπίζω ότι μπορεί να απαντηθεί. Επειδή για την ώρα μαθαίνω ότι όλοι λένε «Α, ο άλλος πρέπει να αρχίσει». Η χώρα μέλος λέει «Όχι, να κάνει την αρχή η Ευρώπη». Η Ευρώπη λέει όχι, να, να καταθέσει αίτηση η χώρα μέλος, κάθε χώρα μέλος. Ποιος είναι αρμόδιος, αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι δηλαδή, ποιος μπορεί να προκαλέσει την λήψη απόφασης. Μπορεί κάποιος να μου δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση, θα σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων. Ποιος μπορεί λοιπόν να δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα. Είναι σημαντική η ερώτηση αυτή. Το ότι καμία χώρα μέλος δεν έχει ζητήσει να αλλάξει, αυτό δεν με εκπλήσει πολύ, διότι σημαίνει και κάποια προσπάθεια. Δεν σημαίνει όμως ότι είναι λάθος η ιδέα της κατάργησης της ελληνικής ώρας. Ε, yes, I will... Ευχαριστώ πολύ. Μία ακόμα ερώτηση θα ακούσουμε και μετά θα ακούσουμε τις πρώτες απαντήσεις και στη συνέχεια θα ακούσουμε και άλλες ερωτήσεις. Ο κύριος Στεχόφσκι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ε, αρχίσατε αυτή τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι εδώ αρκετά εξέχουσες προσωπικότητες ε, που ε, τους ενδιαφέρει αυτή η συζήτηση και θα ήθελα να πω επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχολούμαστε με θέματα που απασχολούν τους συμπολίτε μας. Εδώ και 6 χρόνια ασχολούμαι με αυτό το θέμα και έχω λάβει εκατοντάδες ε, γράμματα, έχω διαβάσει δεκάδες μελέτες σε σχέση με το θέμα αυτό. Δεν θα μπω σε κριτική της Οδηγίας Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής δεν θα μιλήσω για όλα, απλώς θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες έρευνες που δεν αναφέρθηκαν ακόμα. Το 2008 στο ε, New England of Medicine ε, παρουσιάστηκαν κάποιες μελέτες οι οποίες κατέδειξαν ότι οι, τις τρεις πρώτες εβδομάδες μετά την αλλαγή της ώρας από τη χειμερινή στη θερινή, ο αριθμός των καρδιακών προσφολών, των εμφραγμάτων αυξήθηκε. Μία ακόμη μελέτη του 2007 αυτή τη φορά, στο Science Daily, αναφέρει ότι ο άνθρωπος αντιδρά στην αλλαγή. Υπάρχουν λοιπόν νέες μελέτες ε, οι οποίες δείχνουν πόσο κακή είναι αυτή η αλλαγή της ώρας από χειμερινή σε θερινή και από θερινή σε χειμερινή στη συνέχεια. Υπάρχουν και άλλες μελέτες ε, πιο πρόσφατες Μήπως αυτές οι μελέτες είναι αντικείμενο, είναι αντίδραση στις δικές μας ε, συζητήσεις. Το θέμα, για παράδειγμα, της, ε, των συνεπειών στο βιολογικό μας ρυθμό. Υπήρξε μία ακόμη μελέτη βάσει της οποίας ότι αυξάνονται μία εβδομάδα μετά την αλλαγή της ώρας και τα ποσοστά των αυτοκτονιών. 5 με 7% μάλιστα. Αυτό είναι το ποσοστό την πρώτη εβδομάδα μετά την αλλαγή της ώρας. Κάτι ακόμη, ο αριθμός των ατυχημάτων. Οδικών. Γιατί μιλήσαμε για τις μεταφορές. Το ερώτημα που θέτω εγώ είναι το εξής. Πώς θα αντιδράσουμε σε όλες αυτές τις μελέτες στο ε, Sleek Medicine για παράδειγμα που λέει ότι αυξάνεται ο αριθμός των οδικών ατυχημάτων κατά 8% την εβδομάδα μετά την αλλαγή της ώρας. Ε, στη Σουηδία 11% είναι αυτό το ποσοστό. Είναι κάποια αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι υπάρχει ή όχι φως έχει κάποιες συνέπειες. Μπορούμε να μιλήσουμε για μια συστηματική αύξηση από τη μία χρονιά στην άλλη του αριθμού των ανθρώπων που είναι θύματα ενός οδικού ατυχήματος. Είναι στοιχεία σημαντικά τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να εξετάσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω από τους δύο πρώτους προσκεκλημένους μας να απαντήσουν τις ερωτήσεις που τους ετέθησαν. Κύριε, εσείς πρώτοι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Όπως είπατε βεβαίως, ε, είναι ένα θέμα συναρπαστικό και κάθε φορά ε, που το συζητάμε αυτό το θέμα της θερινής ώρας, όλα αυτά τα παράπονα ε, που, που αναφέρατε εσείς είναι παράπονα που τα ακούμε κι εμείς από το περιβάλλον μας. Από, απόψε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής όμως που πρέπει να χειριστεί την εναρμόνιση των ενδεχόμενων συνεπειών στην εσωτερική αγορά φοβούμε ότι το μόνο που μπορούμε να πούμε για την ώρα είναι καταρχάς θα μπορούσαμε να ε, συζητήσουμε κατά πόσο θα καταργήσουμε ή όχι αυτήν την οδηγία. Αν την καταργήσουμε τι θα κάνουμε αν ένα ε, κράτος μέλος αποφασίσει να διατηρήσει την αλλαγή της ώρας. Τότε ξαναπάμε προς τα πίσω. Η πρώτη λύση θα έπρεπε να είναι ε, ε, στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς θα μπορούσαμε να απαγορεύσουμε σε όλα τα κράτη-μέλη την αλλαγή της ώρας από χειμερινή σε θερινή. Αλλά μέχρι τώρα τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει, ζητήσει, δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από τα κράτη-μέλη, από κανένα κράτος μέλος. Ε, τα διάφορα παράπονα που ακούσαμε ε, δεν ήταν εκατοντάδες ή χιλιάδες, ε, ήταν πολύ λίγα και προέρχονταν από κάποιους πολίτες, ε, μία ή δύο οργανώσεις στην Ευρώπη. Οι επιχειρήσεις δεν αναστατώνονται πάρα πολύ από την αλλαγή της ώρας, αντιθέτως θέλουν ε, ένα μακροχρόνιο προγραμματισμό σαφή για το πότε θα αλλάξουν τα πράγματα αν αλλάξουν. Οπότε εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είμαστε βέβαιοι για το τι θα συμβεί. Θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών ή όχι. Στο, συμβούλιο, στο Κοινοβούλιο θα υπάρξει ε, ε, συμφωνία. Όπως είπα, από ε, θεσμικής απόψεως δεν έχουμε πολλά περιθώρια ελιγμών γιατί η απόφαση ε, για την ώρα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα ε, του κάθε κράτους μέλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να απαντήσω το ερώτημα για το χρονοδιάγραμμα των ε, μεταφορών των οράνιων τρένων. Δεν είμαι βέβαιος ότι κατάλαβα πάρα πολύ καλά. Θα σας πω όμως είναι εύκολο να βρούμε νούμερα που θα μπορέσουν να αιτιολογήσουν αυτό που θέλουμε να πούμε. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα για την αύξηση των ατυχημάτων το φθινόπωρο και τη μείωση το καλοκαίρι, για τα οδικά ατυχήματα πιστεύουμε ότι θα συνέβαιναν ούτω ή άλλω, γιατί ο αριθμό των ορών με φω μειώνεται. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο όμω με το φω, μπορεί να έχει να κάνει με την εποχιακή διακύμανση ούτω ή άλλω. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή να το, αποδώσουμε υποχρεωτικά στην αλλαγή της χώρας και στην έλλειψη φωτό... φωτός. Νομίζω ότι αυτά θα μπορούσα να πω σε σχέση με τις ερωτήσεις που άκουσα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Άλλες ερωτήσεις, Μπέκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Ευχαριστώ και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τον εμπειρογνώμονα που μας παρέχουν τις πληροφορίες αυτές. Για μένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ωστόσο, το ξεκαθαρίζω, έχει το χρέος να αναλάβει πρωτοβουλία. Το πώς μετά, τι συνέχεια θα δοθεί στο νομοθετικό χώρο είναι άλλη υπόθεση. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει την ευθύνη να αναλάβει πρωτοβουλία. Δεύτερο, όπως και ο συνάδελφός μου, θεωρώ ότι δεν υπάρχουν επιστημονικά θεμελιωμένες μακροπρόθεσμες μελέτες. Υποθέτω και ισχυρίζομαι επίσης ότι και όλες οι μελέτες εκείνες που μιλούν δυστυχώς για πολλούς νεκρούς και ατυχήματα κτλ δεν έχουν εξεταστεί με την ίδια σοβαρότητα. Μπορείτε να με διορθώσετε. Γνωρίζουμε όμως ότι από μαθητές μέχρι ηλικιωμένους γνωρίζουμε από πολλές μελέτες ότι για όλες τις ηλικίε προκύπτουν σοβαρές δυσκολίες. Εκεί δεν βλέπω να έχει γίνει καμιά αξιολόγηση. Δεύτερο, θεωρώ ότι οι επιχειρήσεις δεν θα υποστούν απολύτως καμιά ζημιά από μια ενδεχόμενη κατάργηση επιχειρήσεις είναι αρκετά εύκαμπτες και ευέλικτες για να αντιμετωπίσουν μια τέτοια αλλαγή. Τρίτο, δεν θα πρέπει να τίθεται το ερώτημα εγκατάλειψης της θερινής ώρας. Θα πρέπει να τεθεί το ερώτημα της αλλαγής της ώρας καθε αυτήν. Ίσως αργότερα κάποιος να προβάλλει το επιχείρημα για την διατήρηση, όλο το έτος εννοεί, της θερινής ώρας. Δεν το ξέρω ίσως. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι η αξιολόγηση του ερωτήματος γιατί χρειάζεται η αλλαγή της ώρας. Εάν δεν υπάρχουν αξιοσημείωτα ωφέλη από άποψη εξοικονόμησης ενέργειας. Και αν δεν υπάρχουν και συγκεκριμένες εμπειρίες που να έχουν μετρηθεί για τις μεταφορές. Αυτά είναι λοιπόν δύο ξεχωριστά θέματα αν δεν υπάρχει ο χρόνος, τότε την απόφαση για το θέμα αυτό θα πρέπει, η απόφαση αυτή θα πρέπει να αναβληθεί. Εδώ μιλούμε για χιλιάδες ανθρώπων και για δισεκατομμύρια ευρώ. Βρίζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τις τρεις κοινοβουλευτικές επιτροπές που οργάνωσαν την ακρόαση. Ο συντονιστής του Λαϊκού Κόμματος είχα ζητήσει μάλιστα να λάβει η... να συμμετάσχει και η Επιτροπή που ασχολείται με τη δημόσια υγεία. Δυστυχώ οι άλλοι συνάδελφοί μου δεν υποστήριξαν την ε, πρότασή μου αυτή. Πάντω χαίρομαι που γίνεται η ακρόαση και το βρίσκω πολύ σημαντικό. Όπω είπαν και άλλοι συνάδελφοί μου, τα υποστηρίζω και εγώ αυτά, και επανέρχομαι. Η εκπρόσωπο τη Κομισιόν λέει κάτι που ακούμε εδώ και μήνε και χρόνια μάλιστα, ότι καμιά χώρα μέλο δεν, δεν έχει υποβάλει το αίτημα κατάργησης της θερινής ώρας. Αυτό όμως είναι και ένας απλός κύκλος. Μία χώρα μέλος δεν αρκεί. Θα πρέπει να διεξαχθεί μια πανευρωπαϊκή συζήτηση. Γι' αυτό και κάνω μια ερώτηση και παρακαλώ μου δώστε μια προσεκτική αν θέλετε απάντηση που να λαμβάνει όμως υπόψη τη σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν δηλαδή το Κοινοβούλιο αναλάβει έκθεση πρωτοβουλίας και ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αυτήν να αναλάβει την πρωτοβουλία, θα το πράξετε. Μπορεί κανείς να συνοηθεί τότε με τις χώρες μέλη. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν υπάρχει πολιτική βούληση εκ μέρους της εμφανίζεται αρκετά δημιουργική και κάνει προτάσεις. Μην έρθετε τώρα να μου πείτε ότι αυτή τη φορά δεν γίνεται. Δώστε μου αν θέλετε μια απάντηση που να λαμβάνει υπόψη τη σχέση μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ η κυρία Χαουτάλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω και να στηρίξω όλα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι μέχρι τώρα. Σε σχέση με αυτά που μας είπε ο εμπειρογνώμονας ε, για την οδική ασφάλεια, έχω να πω ότι αυτό που πιστεύω ότι ακούσαμε είναι ότι ε, στην καλύτερη των περιπτώσεων αυτή η εξοικονόμηση ε, φωτός της ημέρας ε, είναι οπωσδήποτε ε, άνισα κατανεμημένη. Εμείς έχουμε, υποφέρουμε από την έλλειψη του φωτός της ημέρας. Για φανταστείτε Φιλανδία το Δεκέμβριο, πόσο λίγο φως ημέρας βλέπουμε. Εν πάση περιπτώσει υπάρχουν και στοιχεία τα οποία είναι αντικρουόμενα. Λέμε ωραία αυτό είναι καλό για την οδική ασφάλεια, αλλά ας πούμε στη Γερμανία επειδή ακριβώς έχουν περισσότερη μέρα ε, που διαρκεί περισσότερο ημέρα, θα βγουν περισσότερο άρα ε, κινδυνεύουν από περισσότερα ε, οδικά ατυχήματα. Το θέμα είναι να καταλάβουμε την ε, φιλοσοφία της ε, ε, Κομισιόν. Τώρα με τη νέα Κομισιόν Γιούνκερ, ε, ο Αντιπρόεδρος Τίμερμαντς μας λέει συνέχεια όλα πρέπει να έχουν προστιθέμενη αξία. Τούτο εδώ τώρα το νομοθέτημα τι προστιθέμενη αξία έχει. Εγώ αμφιβάλλω αν έχει οποιαδήποτε. Επομένως θεωρούμε ότι θα πρέπει αυτή η οδηγία, ε, ότι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να αποσυρθεί σαν μια σημαντική πρωτοβουλία στα πλαίσια του προγράμματος REFIT. Εγώ είπα κάποια στιγμή στο facebook ότι στα πλαίσια του Refit θα πρέπει να καταργηθεί η οδηγία για τη θερινή ώρα και δεν ξέρω κι εγώ πόσα likes πήρα, χιλιάδες. Και όσον αφορά τώρα αυτό που είπατε σχετικά με τις επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, τι εννοείτε, ότι δεν μπορούμε και δεν πρέπει να, να, να προτείνουμε καμία ε, αλλαγή στην νομοθεσία. Δεν νομίζω ότι έχετε δίκιο. Ο κύριος Λίζε πολύ σωστά είπε ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να βοηθήσει και την Κομισιόν όσον αφορά κάποια συμπεράσματα και άλλωστε έχουμε και εμείς ε, το ε, ανεπίσημο ε, δικαίωμα πρωτοβουλίας. Εν πάση περιπτώσει εμείς εκπροσωπούμε ανθρώπους οι οποίοι φαίνεται ότι ενοχλούνται από αυτήν την οδηγία και νομίζω ότι στην ουσία αυτό που είπε ο άλλος συνάδελφος είναι σημαντικό αυτό που αλλάζουμε συνέχεια τα ρολόγια. Ε, και όταν αλλάζουμε την ώρα έχουμε την αίσθηση το Μάρτιο ότι φέρνουμε το χειμώνα και τον, αυτό ότι φέρνουμε το καλοκαίρι. Γιατί να τα αλλάζουμε τα ρολόγια μας. Νομίζω ότι θα πρέπει να ρωτήσω τώρα τους έγκριτους καλεσμένους μας εάν θέλουν να απαντήσουν. Παρακαλώ κυρία μου. Κοιτάξτε. Συγχωρέστε με εάν Ε, είπα κάτι λανθασμένο. Η Κομισιόν όντω έχει δυνατότητα ε, τέτοια πρωτοβουλία, αλλά φυσικά και το Κοινοβούλιο μπορεί να, κάνει τέτοιου είδους, να αναλάβει τέτοιου είδου πρωτοβουλία. Όπως σας είπα και προηγουμένως, για την ώρα εμείς σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχουμε λάβει επίσημο αίτημα από πλευράς ε, ε, κάποιας χώρας. Ναι, έχουμε δυνατότητα ε, να δράσουμε από μόνοι μας, αλλά, αλλά πριν ε, παρουσιάσουμε ε, οποιασδήποτε προτάσεις ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να παρουσιάσουμε στοιχεία και καλά στοιχεία, γερά στοιχεία μέσα από μελέτες αντικτύπου. στα πλαίσια της ε, καλύτερης νομοθέτησης ε, οτιδήποτε μπορούμε να το κάνουμε, είτε να κάνουμε νέα πρόταση, είτε να αποσύρουμε την υφιστάμενη, ε, είναι, εξακολουθεί να είναι δυνατότητα. Αλλά βέβαια, εάν αποσύρουμε την υφιστάμενη, τότε παραμένουμε στο πρόβλημα το οποίο ανέφερα προηγουμένως. Εάν μία, δύο, τρεις, πέντε χώρες από τις 28 αποφασίσουν ότι διατηρούν αυτή την αλλαγή ώρα, δεν νομίζω ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα οι επιχειρήσεις. Ενδεχομένως με μονομένες επιχειρήσεις στην Α ή στη Β δεδομένη χώρα ίσως δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα, αλλά γενικότερα οι πολλοί κλάδοι θα έχουν πρόβλημα. Ναι, δεν λέω ότι δεν έχουμε δικαίωμα ή δυνατότητα πρωτοβουλίας, ωστόσο αυτό που λέω είναι ότι τα στοιχεία και οι διαμαρτυρίες που έχουμε ε, λάβει μέχρι τώρα δεν μας οδηγούν σε μια ανάγκη απόσυρσης ε, της οδηγίας. Αντιθέτως, εγώ ενθαρρύνω το Κοινοβούλιο να προχωρήσει σε συγκεκριμένες δράσεις ε, οι οποίες θα μας οδηγήσουν στο να ξανασκεφτούμε το, το ζήτημα αυτό. Αυτό θα μπορούσε πραγματικά να αποτελέσει μια πολύ καλή πρωτοβουλία των εξονόματος των πολιτών η Κομισιόν δεν λέει ότι τα επόμενα 100 χρόνια δεν πρέπει να αλλάξει τίποτα. Λέει ότι στα πλαίσια της καλύτερης νομοθέτησης ό,τι μας προτείνεται θα το μελετήσουμε εντελεχώς. Ευχαριστώ. Ναι, θα ήθελα να επανέλθω και εγώ ίσως ξεκινώντας από το τελευταίο σημείο. Όντως είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ε, ότι δεν είναι ίδια η επίπτωση σε ολόκληρη την Ευρώπη και ότι κάποιοι έχουν πλεονεκτήματα και ωφέλη και άλλοι αντιστοίχω ε, ζημιώνονται. Ε, εγώ όμως πιστεύω ότι όσον αφορά την μείωση των οδικών ατυχημάτων πιστεύω ότι ε, το, το όφελος είναι σημαντικό. Είναι δύσκολο βέβαια να δώσουμε συγκεκριμένο αριθμό και όντως σε κάποιες περιπτώσεις ίσως μπορεί να υπάρχουν ε, κάποια, ε, ε, κάποια στοιχεία συνοδευτικά τα οποία δεν είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό ε, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούμε να πούμε ότι ε, θα απαγορεύσουμε πούμε, τα νυχτερινά ταξίδια γιατί μπορεί να προκληθούν τότε περισσότερα ε, ατυχήματα. Εγώ νομίζω ότι σε γενικέ γραμμέ, βλέποντα τα υπέρ και τα κατά, βλέποντα τα ωφέλη και τι τις νομίζω ότι τα ωφέλη είναι περισσότερα. Ε, είναι γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, αλλά ίσως, αυτό το ίσως θα πρέπει να θυσιάσουν κάτι στον βωμό του κοινού καλού. Ναι, νομίζω ότι ενδεχομένως ορισμένοι θα πρέπει να θυσιάσουν κάτι και ίσως αυτό πράγματι δεν είναι καθόλου καλή, εύκολη και ευχάριστη απόφαση. Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώθηκε λοιπόν ε, ερώτηση μάλλον την κυρία Κάουφμαν. Ευχαριστώ. Εγώ έχω μια ερώτηση αντίθετα με αυτά που είπαν οι μέχρι τώρα ραλίσαντες. Εγώ δεν θα κρίνω την θερινή ώρα είναι καλή ή κακή, αλλά ακρόαση κάνουμε εδώ. Επιθυμώ να ρωτήσω λοιπόν τον εμπειρογνώμονα εκ Μεγάλης Βρετανίας, γιατί εμένα με απασχολεί αυτή η σχέση μεταξύ του αριθμού των νεκρών από οδικά ατυχήματα και της θερινής ώρας, όπως την παρουσίασε θεωρεί ότι είναι ασφαλώς επιστημονικά θεμελιωμένη η αναλογία αυτή, η διασύνδεση αυτή. Διότι βέβαια μπορεί να υπάρχουν και άλλα αίτια για τα οδικά ατυχήματα, π.χ. η τεχνική κατάσταση των οχημάτων, το εάν ο οδηγός ε, τελεί ε, σε κατάσταση μέθηση όχι. Και βέβαια παίζει ρόλο ο αριθμός των συμμετεχόντων στην κυκλοφορία. Γνωρίζουμε όμως ότι ο αριθμός των αυτοκινήτων έχει αυξηθεί εκθετικά στους δρόμους μας και δεν με εκπλήσει ότι σε περιόδους, σε ώρες δηλαδή κυκλοφοριακής εχμής ασφαλώς τα ατυχήματα είναι και περισσότερα. Αυτό δεν νομίζω όμως ότι έχει σχέση τόσο πολύ με τη θερινή ώρα όσο με το ότι είναι όντως κυκλοφοριακή αιχμή. Μήπως μπορείτε να πείτε δύο λόγια για αυτά τα πράγματα. Αν δηλαδή υπάρχει μια πραγματική άμεση συνάφεια ανάμεσα στον αριθμό των ατυχημάτων και βεβαίως των νεκρών από ατυχήματα, ε, από αυτοκινητικά δηλαδή δυστυχήματα και ε, την ηθερινή ώρα. Η κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα τσεχικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον συμφωνώ με όλους όσους ε, θα ζητούσαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονηθεί μία μελέτη σε σχέση με τον αντίκτυπο της αλλαγής, της κατάργησης αλλαγής ώρας. Ο γερουσιαστής ε, Σίλε δεν ε, ήξερε ακριβώς ε, τι συνένεση θα υπήρξε θα υπήρχε γι' αυτό. Η ιδέα είναι να ε, απλοποιηθεί η κατάσταση και να καταργηθούν οι άχρηστες αλλαγές ώρας. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μία τεχνοκρατική προσέγγιση, εντελώς επιστημονική, εντελώς αντικειμενική, σε σχέση με το ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος ε, της κατάργησης αλλαγής της ώρας. Θα έπρεπε Προφανώς να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη, να συμφωνήσει και το Κοινοβούλιο. Έχει καταλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία. Εγώ ευχαρίστως να συντάξω μία γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας της ε, να εκπονήσει ε, μελέτη αντικτύπου και ενδεχομένως να τροποποιήσει και τη σχετική οδηγία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολύτιμο ρόλο να διαδραματίσει γιατί ακούμε τι μας λένε στις περιφέρειές μας οι συμπολίτες μας. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε τις απαντήσεις. Έχετε το λόγο. Ναι, όσον αφορά τη μελέτη αντικτύπου, για να δούμε τον αντίκτυπο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα μπορούσε να εκπονήσει μία μελέτη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία άλλη, ώστε να υπάρχει έτσι, μια ουδέτερη μια ουδετερη αντιμετωπιση των πραγμάτων. Υπάρχει όμως ακόμη το ζήτημα ε, του προϋπολογισμού για τις προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker. Και για την ώρα, η θερινή ώρα δεν ε, εγγράφεται μεταξύ των προτεραιοτήτων αυτών, αλλά κατόπιν ετήματος ενός από τους ε, συνομοθέτες μας ε, και αν υπάρχει δυνατότητα στον προϋπολογισμό, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Ναι, απαντώντας την πρώτη ερώτηση, θα ήθελα να πω όλα τα ατυχήματα είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων, ε, είτε είναι το όχημα, είτε είναι το φως, ε, είτε είναι κουρασμένος ο οδηγός, ε, όταν γίνεται υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Τα ατυχήματα γίνονται όταν πολλοί παράγοντες υπησέρχονται παράλληλα. Δεν μπορούμε να πούμε αυτό το ατύχημα έγινε λόγω της έλλειψης φωτός και δεν θα είχε συμβεί αν υπήρχε περισσότερο φως. Αλλά μπορούμε να δούμε μία απότομη αύξηση στην αλλαγή στην αύξηση των ε, ατυχημάτων ε, όταν είναι σκοτάδι σε σχέση με το όταν υπάρχει φως. Ε, κάποια ατυχήματα σίγουρα οφείλονται σε αυτό το λόγο. ο, οι συνολικοί αριθμοί δείχνουν ότι υπάρχει μία σημαντική διαφορά. Εμείς τώρα προσπαθούσαμε αυτό να το παρουσιάσουμε κάπως. Εσείς μιλήσατε για τον αριθμό των ατυχημάτων ε, ανά ε, χιλιόμετρο. Ναι, θα μπορούσαμε να, προσθε... να, να, να ε, συγκρίνουμε δύο ε, ε, παράλληλους αριθμούς για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο από έναν αριθμό και μόνο ατυχημάτων να πούμε «Α, αυτό το ατύχημα οφείλεται στο σκοτάδι, αυτό το ατύχημα δεν οφείλεται». Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι ε, να πούμε ε, κατά πόσο, τουλάχιστον εν μέρη, όταν υπάρχει περισσότερο φως γίνονται λιγότερα ατυχήματα. Ελπίζω να απάντησα στην ερώτησή σας. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο τμήμα της ακρόασής μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους προσκεκλημένους μας τους δύο πρώτους προσκεκλημένους μας ε, για αυτό το πολύ αισιόδοξο μήνυμα ότι έχουμε ισχυρούς συμμάχους ε, η Επίτροπος Μπιενκόφσκα, ε, τη υπεύθυνη για την εσωτερική αγορά, μας είπε ότι είναι υπέρ της κατάργησης της αλλαγής της ώρας. Είναι λοιπόν σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουμε τέτοιους συμμάχους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερο τμήμα της συνεδρίασής μας, η καθηγήτρια Μάρτα Μέρουφ από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου και από το τμήμα της ιατρικής ψυχολογίας. Έχετε το λόγο. Κύριε Σφοβόντα, κύριε Μπούζεκ, κυρίες και κύριοι, Ευρωβουλευτές. σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να είμαι εδώ σήμερα και να είμαι με αυτή τη σημαντική συζήτηση για το τι να κάνουμε με τη θερινή ώρα. Ακούσατε για τον τουρισμό, ε, για την οικονομία, ε, για την ε, κυκλοφορία. Θα προσπαθήσω και εγώ να σας πω κάποια πιο επιστημονικά στοιχεία. Εγώ προέρχομαι από το τμήμα ιατρική ψυχολογία του Πανεπιστημίου του Μονάχου εγώ δεν εκπροσωπώ τόσο το, τα, την, ε, τον εαυτό μου όσο την, ολόκληρη την εργασία για το θέμα της ε, χρονοβιολογίας. Ο συνάδελφος επίσης προέρχεται από το τμήμα ιατρικής ψυχολογίας. Θα προσπαθήσω να ε, σας, παρουσιάσω κάπως γρήγορα ε, τον τομέα μου, να σας παρουσιάσω ε, ορισμένα πράγματα. Σκεφτείτε λίγο ε, όλους όσους ζουν μαζί σας όταν, και κυρίως το πότε κοιμούνται σε σχέση με το πότε κοιμάστε εσείς. Οι περισσότεροι θα αναγνωρίσετε ότι κάποιοι άλλοι στο σπίτι σας κοιμούνται νωρίτερα ή αργότερα από εσά, οι έφηβοι κοιμούνται πολύ αργότερα, τα μικρότερα παιδιά πολύ νωρίτερα, ε, κάθε ένας έχει μια συγκεκριμένη προτίμηση για, το χρονικό, ε, για τη χρονική στιγμή στην οποία θα κινηθεί. Αυτή όμως η προτίμηση δεν είναι τόσο ε, προτίμηση, δεν επιλέγει κανείς το χρονότυπό του και την ώρα του ύπνου, γιατί ελέγχεται από το βιολογικό του ρολόι και το βιολογικό ρολόι προγραμματίζεται ε, στα γονίδια σας. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Δεύτερο σημείο ο χρονισμός ε, της, ε, του ύπνου είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου, γιατί το βιολογικό ε, ρολόι μας καθορίζει και τις ορμόνες μας και τη συμπεριφορά μας, τις επιδόσεις μας, το γνωστικό μας το και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε είναι να προσαρμοστούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρξει όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του οργανισμού σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Τρίτη έννοια, το κυρκάδιο ε, ρολόι παίρνει ε, σήματα συνέχεια από το περιβάλλον, ε, από το φως και από το σκότος. Αυτά τα δύο μαζί χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή του βιολογικού μας ρολογιού. Ο αντίκτυπος του φωτός στο βιολογικό ρολόι μας είναι τόσο ισχυρός που αν ζει κανείς στην ανατολική πλευρά της ζώνης ώρας, ε, ε ξυπνάει κανείς πιο νωρίς γιατί ανατέλει ο ήλιος νωρίτερα. Ο αντίκτυπος του φωτός είναι τόσο ισχυρός που λιγότερο φως ε, κατά τη διάρκεια της ημέρας ε, σημαίνει ότι εσείς γίνεστε ε, πιο νυχτερινός τύπος. Είναι τόσο ισχυρός λοιπόν ο αντίκτυπος του φωτός στο βιολογικό ρολόι που αν κανείς εκτίθεται περισσότερο σε φως το βράδυ τότε το πρωί, από ότι το πρωί τότε θα γίνει κανείς πιο νυχτερινός τύπος σε σχέση με κάποιον άλλον. το ρολόι που επηρεάζει ε, το ωράριο εργασίας μας για παράδειγμα, ε, αν συνείδε πλήρως με το ε, βιολογικό μας ρολόι δεν θα χρειαζόμασταν ξυπνητήρια. Όμως 80% του πληθυσμού χρησιμοποιεί ε, ξυπνητήρι στις ε, ε, εργάσιμες ημέρες. Γιατί είναι μεγάλο αυτό το ποσοστό? Γιατί υπάρχει ένα κοινωνικό πρόγραμμα, υπάρχουν τα ωράρια της δουλειάς και του σχολείου που σημαίνει ότι πρέπει να ξυπνήσουμε νωρί. Τάση λιγότερου φωτό στο περιβάλλον μας, κάτι το οποίο σημαίνει ότι γινόμαστε πιο νυχτερινοί τύποι και υπάρχει και το θέμα βέβαια της θερινής ώρας που πιέζει ακόμη περισσότερο το βιολογικό μας ρολόι. Όταν ε, χρησιμοποιούμε ένα ξυπνητήρι, σημαίνει, τι σημαίνει, ότι τις ημέρες που δουλεύουμε πρέπει να ξυπνήσουμε μια συγκεκριμένη ώρα ε, και ξυπνάμε πολύ νωρίτερα από την ώρα που θα μας ξύπνε και το βιολογικό μας ρολόι. Επομένως, ε, ο ύπνος μας μειώνεται και δεν είναι, δεν είναι η στιγμή που κοιμόμαστε δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Όσον αφορά τώρα το jet lag για παράδειγμα, όταν κανείς ε, ταξιδεύει σε μεγάλες αποστάσεις, ε, το ίδιο μπορεί να επιτευχθεί με ε, την έλλειψη ύπνου. Είναι το κοινωνικό jet lag που προκύπτει από την ανάγκη του να πάμε σχολείο ή να δουλέψουμε και να ξυπνήσουμε νωρί. Αν το jet lag δεν συμβαίνει πολύ συχνά, δεν υπάρχουν σοβαρές συνέπειες, όμως το κοινωνικό jet lag είναι μία συνεχής κατάσταση κάθε εβδομάδα που συνεχίζεται για όλη τη διάρκεια της καριέρας μας ε, και έτσι δημιουργείται μια χρόνια συμπεριφορά. Μερικές φορές δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι έλλειψη ύπνου που σημαίνει χειρότερες επιδόσεις, κακή κρίση και αλλαγές στην προσωπικότητα όπως για παράδειγμα μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες άλλοι, σε άλλες συνέπειες του κοινωνικού jet lag έχει να, έχουν να κάνει με την ε, έλλειψη ύπνου ή με το ότι είναι κανείς ξύπνιος και δραστήριος στη λάθος χρονική στιγμή. Αυτό έχει επίσης αμέσως σχέση με την ε, κατανάλωση νοπνευματοδών ποτών, το κάπνισμα, ε, την καφεΐνη, την υπερβολική χρήση της καφεΐνης την κατάθλιψη, μεγάλα προβλήματα του 21ου αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγάλη αύξηση κάποιων συγκεκριμένων συμπεριφορών που οφείλεται στο κοινωνικό jet lag. Περισσότερο κοινωνικό jet lag, περισσότερη παχυσαρκία για παράδειγμα ή περισσότερη κατάθλιψη. Αυτά είναι στοιχεία που είναι απαραίτητα για να καταλάβουμε πώς επηρεάζει η αλλαγή της ώρας ε, την, τον οργανισμό μας. Η θερινή ώρα ε, σημαίνει ότι το κοινωνικό μας ρολόι πάει πίσω μία ώρα και το χειμώνα αυτό αλλάζει. Όμως το, ο αντίκτυπος του φωτός στο κοινωνικό μας, στο βιολογικό μας ρολό είναι τόσο σημαντικός που ουσιαστικά ε, δεν ορίζεται πια από το κοινωνικό μας ε, κομμάτι αλλά από το βιολογικό μας κομμάτι το πότε θα ξυπνήσουμε. Ε, ξυπνάμε λοιπόν πολύ νωρίτερα και το αποτέλεσμα είναι ότι όλο και περισσότερο μεγαλώνει το κοινωνικό jet lag. υπάρχουν πολύ περισσότερες καρδιοπάθειες, ε, εμφράγματα μετά την αλλαγή της ώρας και υπάρχουν και χρόνια συνέπειες. Ε, η μετάβαση στη θερινή ώρα σημαίνει περισσότερο κοινωνικό ε, jet lag, περισσότερα τσιγάρα, περισσότερη παχυσαρκία, περισσότερο διαβήτη τύπου 2, περισσότερη κατάθλιψη. Αυτή είναι, αυτές είναι σύγχρονες επιδημίες που σημαίνουν απώλειες για τον τομέα της ιατρικής περίθαλψης. 1% ε, του ΑΕΠ στην περίπτωση αυτή θα σήμαινε 131 δισεκατομμύρια ευρώ ε, κατέτος μας στοιχίζει αυτό η κατάργηση της αλλαγής της ώρας και η μείωση του κοινωνικού jet lag φυσικά θα μείωνε αυτό το ποσό. Το ποσό μπορεί να φαίνεται πολύ διωγγωμένο, αλλά νομίζω ότι είναι ε, μάλλον ε, μια υποτίμηση της πραγματικότητας, αν λάβουμε υπόψη, για παράδειγμα, ε, την κατάσταση των εφήβων, που είναι οι πιο νυχτερινοί τύποι ε, και οι οποίοι υφίστανται τις περισσότερες συνέπειες της αλλαγής αυτής. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικός και ο ρόλος της εκπαίδευσης ε, και ειδικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόσφατα φάνηκε ότι η νυχτερινή τύπη που είναι η έφηβοι με κοινωνικό jet lag ε, ε, σημαίνει ότι οι επιδόσεις τους είναι χειρότερες σε εξετάσεις που λαμβάνουν χώρα πρωινέ πρωινές ώρες από ό,τι καν γίνονται κάποια στιγμή πιο μετά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό επηρεάζει βέβαια τα πανεπιστήμια και αυτό σημαίνει ότι όποιος μπαίνει στο πανεπιστήμιο είναι αυτός που έχει ένα συγκεκριμένο συγκεκριμένο χρονότυπο. Από απόψεως λοιπόν επιστημονικής προτείνουμε ε, να υπάρξουν λύσεις για το πρόβλημα αυτό, ε, κάτι το οποίο θα σήμαινε αύξηση του φωτός ε, κατά τη διάρκεια της ζωής μας και κατάργηση της αλλαγής της ώρας. Όλα αυτά θα μείωναν το κοινοτικό jet lag στον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you, madam. Σας ευχαριστώ και εγώ κυρία μου. Θα ακούσουμε τώρα τη δεύτερη τοποθέτηση. Δόκτωρ Βέρνερ Βαντεμπράνε από το Πανεπιστήμιο της Αμβέρσας. Έχετε 10 λεπτά κύριε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Από την άποψη της καλύτερης νομοθεσίας έχω τέσσερα σχόλια. Θα αρχίσω με τις οδηγίες. Πρώτα η νομική βάση και η η επεξήγησή της το 1999. και θα έρθω μετά και στην εκ των υστέρων αξιολόγηση του 2007. Τώρα, εισαγωγικά. Ποια είναι η σημασία του evidence-based lawmaking. Χρειάζεται ισορροπία ανάμεσα στην πολιτική διάκριση, δηλαδή στην ευκαιρία. Δυστυχώς ο μιλητής μιλεί με μεγάλη ταχύτητα, είναι αδύνατον να παρακολουθεί. με τα impact assessment το δικαστήριο μπορεί να παρακολουθήσει την αξιολόγηση από τον νομοθέτη περίπλοκων κοινωνικονομικών δικτών. Οι μελέτες επιπτώσεων είναι το βασικό εργαλείο για να εξασφαλίζεται η διατήρηση της αναλογικότητας και της επικουρικότητας, ιδίως για την οδηγία περιθυρινής ώρας Το επεξηγηματικό μνημόνιο έχει τον ίδιο σκοπό να επιτρέψει δηλαδή την επιλογή των νομικών όρων. Πρώτα η νομική βάση για την οδηγία 2084 είναι η διάταξη του άρθρου 114 της Συνθήκης της Λισαβόνας που επιτρέπει την έγκριση μέτρων, κυρίως οδηγιών, για την εναρμόνιση εθνικών μέτρων για να βελτιωθεί η λειτουργία της ενιαίας αγοράς του άρθρου 26 της ίδιας συνθήκης. Το δικαστήριο μπορεί να βρει την εφαρμοσιμότητα της αρχής αυτής πρώτον με την προτεραιότητα του ειδικού νόμου δεύτερο με τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς όταν δεν επαρκούν οι εθνικές διατάξεις και υπάρχει βελτίωση Υπάρχει η υπόθεση Vodafone με μέτρα υπό την ισχύ του άρθρου 95 για την ίδρυση της ε, ενιαίας αγοράς. για την αποφυγή ανταγωνισμού. Αυτά δεν επαρκούν για να επιλεχθεί το άρθρο 95 ως νομική βάση. Ο νομοθέτης μπορεί να προσφύγει σε αυτό, ιδίως όταν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εθνικών κανόνων, τέτοιες που να έρουν τις βασικές ελευθερίες ή να οδηγούν σε σημαντικές στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Αυτά που θεωρεί το δικαστήριο ως ε, διάκριση δεν ερμηνεύονται εύκολα. Η αναλογία μπορεί να υπάρξει από τις συντρέχουσες αρμοδιότητες του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συστήματος, όπου εκεί απαιτείται αναγκαιότητα για την λήψη μέτρου σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο αναμένει λοιπόν από τον Ομοσπονδιακό Νομοθέτη να κάνει μελέτη για τις ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις. Φέρει το βάρος αποδείξεως και σύμφωνα με το Γερμανικό Δικαστήριο πρέπει να υπάρχει σαφήνεια, αποκλεισμός άσχετων στοιχείων και μεθοδολογική συνέχεια. Στην παρούσα περίπτωση της οδηγίας για τη θερινή ώρα, το μνημόνιο φαίνεται να βασίζεται σε διαβούλευση με οικονομικούς φορείς που έχουν ταχθεί υπέρ της εναρμόνισης της θερινής ώρας. Στο παρελθόν αρκούσαν τα επιχείρηματα αυτά για να πιστεί το δικαστήριο για την ε, εφαρμογή του άρθρου 1. Όμως, το επεξηγηματικό μνημόνιο της ε, οδηγίας 2000 για τη βελτίωση της ενιαίας αγοράς δεν φαίνεται επαρκές. Αναλογικότητα και επικουρικότητα. Επικουρικότητα, εδώ υπάρχουν τρία θέματα. Πεδίο εφαρμογής του μέτρου, κόστος και ε, ωφέλεια. Ιδίως για τις επιπτώσεις επιχειρήσεις και άτομα. Εδώ, επειδή η οδηγία εναρμονίζει εθνικό δίκαιο, είναι και το λιγότερο δυστικό μέτρο. Η αναλογικότητα επιτρέπει και την νομοθεσία σε βάση evidence, αλλά δεν είναι απόλυτα πιστικά τα επιχειρήματα. Βασίζεται σε ανεξάρτητη έκθεση τα αποτελέσματα της οποίας δεν είναι αποφασιστικά, όπως έχει δεχθεί στο Memorandum και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδίως για τη Γεωργία, όπου το Memorandum λέει καθαρά ότι δεν μπορούν να συναχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα, το ίδιο για το περιβάλλον. Οι επιπτώσεις της οδηγίας θερινής ώρας είναι δύσκολο να εκτιμηθούν και για, και για την οδική ασφάλεια και ούτω καθεξής φαίνεται ότι οι μεταφορές και ο τουρισμός ήταν οι κύριες αιτίε για την εναρμόνιση. Όσον αφορά τις μεταφορές, η λεπτομερής αξιολόγηση βασίστηκε σε μία μόνο μελέτη από τη Γαλλία το 1996. Το δικαστήριο απαιτεί σε βάθος αξιολόγηση μέτρων και το ίδιο ισχύει και για την ε, Ευρωπαϊκή Νομοθεσία το δικαστήριο μπορεί να εκτελέσει, να μπορεί να αξιολογήσει την αναλογικότητα μόνο στη βάση των στοιχείων προσκομίζει ο νομοθέτης. E Όσον αφορά τώρα την επικουρικότητα, έτσι όπως ε, αναφέρεται στο σχετικό άρθρο της Συνθήκης Λειτουργίας, αναφέρεται ότι στην, ε, ε, στο επεξηγηματικό μνημόνιο παρέχονται ε, σαφείς επεξηγήσεις, οι οποίες σχετίζονται και με τα όσα ανέφερα ήδη για την παράγραφο 4.1. Ωστόσο, παρα, ωστόσο καταδεικνύει τους μη πιστικούς λόγους και την μη ικανοποιητική αιτιολόγηση για οποιοδήποτε απόφαση έχει και ε, άλλωστε και στην υπόθεση Vodafone ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρει ότι ενδεχομένως ε, το στοιχείο αυτό θα, θα ε, αποβεί σημαντικότατο. Έχω και άλλα στοιχεία για την Vodafone αν θέλετε, μπορώ να σας τα δώσω. Ε, όσον αφορά την ε, οδηγία για τη θερινή ώρα, καμία, ε, κανένα από τα στοιχεία και τις επεξηγηματικές σημειώσεις δεν απαντά στα ερωτήματα τα οποία αφενός αναφέρονται στην διεθνική και διακρατική πλευρά του πράγματος και από την άλλη πλευρά πρέπει να πω ότι ούτε στο επεξηγηματικό μνημόνιο, explanatory memorandum, δεν λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία απόκληση επιχειρήσεις τα οποία υφίσταντο ακόμα και πριν από την πρώτη οδηγία. Βεβαίως το επεξηγηματικό μνημόνιο αναφέρεται ε, στην αντίθεση μίας χώρας μέλη προστιθέμενη αξία. Στην προκείμενη περίπτωση η προστιθέμενη αξία εξαντλείται στην απλή εναρμόνιση και οι ε, ε, πρόσφατες αποφάσεις του δικαστηρίου αλλά και η αξιολόγηση αντικτύπου δεν μας οδηγούν σε ε, ικανά συμπεράσματα. Τώρα, για να τελειώσω μπορώ να σας πω ότι η οδηγία της θερινής ώρας δεν αιτιολογείται από την προσπάθεια της Επιτροπής για καλύτερη νομοθέτηση. Επίσης, η επιλογή νομικής βάσης αναλογικής αλλά και επικουρικότητας δεν μας πείθουν. Αυτά ήθελα να σας πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you uh, Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Μετά από αυτές τις δύο παρεμβάσεις έχετε ε, ως ε, μέλη ε, των Επιτροπών την δυνατότητα να υποβάλλετε ερωτήματα στους έγκριτους ομιλητές. Κύριε Μπέκερ. Μπέκερ, θα είμαι σύντομος. Στην βάση των δύο αυτών παρεμβάσεων θεωρώ ότι δικαιωνόμαστε με την έννοια ότι απαιτείται πλέον επιστημονική αξιολόγηση του status quo. Τώρα, δεν προκαταλαμβάνω το αποτέλεσμα. Ευχαρίστως να αφήσω στην άκρη την προσωπική μου προτίμηση, αλλά υπάρχουν λόγοι, τουλάχιστον από αυτά που άκουσα για τη χρονοβιολογική πτυχή που θεμελιώνουν το ότι δεν πρέπει να γίνεται καμιά άσχετη τροποποίηση του χρόνου στη ζωή των ανθρώπων. Ο κύριος Λίζε, ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους δύο παρεμβαίνοντας για την κυρία Μέρου, την καθηγήτρια κυρία Μέρου. Αν κατάλαβα καλά, Αλλιώ να το επαναλάβει και να εξηγήσει γιατί. Αν κατάλαβα καλά, από τη δική σας σκοπιά δεν είναι μόνο η αλλαγή της ώρας δύο φορές το χρόνο και η εβδομάδα που ακολουθεί, αλλά γενικότερα το γεγονός ότι βάζουμε τη θερινή ώρα, διότι αναγκάζει τον κόσμο να ξυπνά νωρίτερα και διότι το βιολογικό ρολόι των περισσότερων δεν το αντέχει. Και με τον τρόπο αυτό αυξάνονται όλες αυτές οι ασθένειες που εξηγήσατε. Αν κατάλαβα καλά, επαναλαμβάνω. Αυτό σημαίνει όμως ότι όχι μόνο δεν πρέπει να προβαίνουμε σε αλλαγή της ώρας, αλλά μάλιστα θα πρέπει να διατηρήσουμε τη χειμερινή ώρα όλο τον χρόνο. Κάτι που μέχρι τώρα δεν έχουν ζητήσει οι πολίτες που έχουν έρθει σε επαφή μαζί μας. Ευχαριστώ κύριε Ρόιλ. Κυρία Καθηγήτρια, θα ήθελα να μάθω αυτά που εξηγήσατε. έχετε ευρεία κάλυψη επιστημονική. Δηλαδή, θέλω να πω, συμφωνούν πολλοί συνάδελφοί σας μαζί σας. Είναι σχετικά. Είναι δηλαδή σχετικά αδιαμφισβήτητη αυτή η θέση που μας παρουσιάσατε. Δεύτερο, έχετε κάποια εξήγηση για ποιο λόγο οι πραγματικές αυτές περιστάσεις, αυτές οι καταστάσεις δηλαδή, λαμβάνονται τόσο λίγο υπόψη στην δράση της πολιτικής αλλά και της κοινωνίας. Όταν για πρώτη φορά εξέτασα το θέμα μετά από έτοιμα πολίτη και εγώ δεν το βρήκα τόσο σημαντικό. Βρήκα το πρόβλημα ενδιαφέρον μεν, αλλά δεν θεώρησα ότι είναι τόσο σημαντικό. Είναι όμως τόσο σημαντικές οι ζημίες στην υγεία. Αυτό είναι μέγα θέμα. Δεύτερο ή μάλλον τρίτο, μπορεί κανείς να ποσοτικοποιήσει ποιος είναι ο αριθμός των ανθρώπων αυτών. Είναι λίγοι άνθρωποι ή είναι ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού που θίγεται. Αυτά θέλω να θέσω με τις ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να απαντήσουν οι εμπειρογνώμονες. Θα ακούσουμε άλλη μια ερώτηση από τον κύριο Λεμπρετόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα τη σημερινή μας ακρόαση και ευχαριστώ όλους όσοι πήραν το λόγο για το θέμα αυτό της, ε, της θερινής ώρας. Ήλιγκο μας προκαλούν όλα αυτά που ακούμε γιατί αναρωτιόμαστε γιατί δημιουργήθηκε αυτή η θερινή ώρα και άρχισε να εφαρμόζεται γιατί ε, τότε ε, γιατί τα επιχειρήματα τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί ε, καταργούνται, ακυρώνονται το ένα μετά το άλλο. Το θέμα της οδικής ασφάλειας, ε, το επιχείρημα αυτό καταπίπτει λόγω της αύξησης των ατυχημάτων. Για το βιορυθμό επίσης τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Είδαμε ότι ο βιορυθμός διαταράσσεται, ότι προκαλεί προβλήματα υγείας, προβλήματα προβλήματα κόπωσης. Ένα άλλο επιχείρημα που ήταν η οικονομία ε, και η εξοικονόμηση γενικά. Εγώ ακούω έναν αριθμό κόστους για το πέρασμα στη θερινή ώρα και αναρωτιέμαι, είπε η κυρία Μερό, ότι το πέρασμα στη θερινή ώρα σύμφωνα με, τις, ε, ε, με, τις, με τους υπολογισμούς της ε, κοστίζει 131 εκατομμύρια την ώρα, την, το έτος, συγγνώμη, δίσετη το έτος, καλά, κατάλαβα καλά Όσον αφορά τώρα την νομική βάση και αυτή η οποία έχει επιλεγεί για το πέρασμα στη θερινή ώρα φαίνεται ότι και αυτή η νομική βάση δεν είναι εξαιρετικά ισχυρή. Γιατί λοιπόν αποφάσισαν οι χώρες να κάνουν αυτό το ε, εγχείρημα. Μήπως απλώς ήθελαν να δείξουν μια κοινή θέση χωρίς καμία αιτιολόγηση και χωρίς καμία ε, αιτία. Πρόεδρος, πριν δώσω το λόγο στους έγκριτους καλεσμένους μας, θα ήθελα και εγώ να πω το εξή. ο κύριος Λεμπρετών φαντάζομαι ξέρει ότι θα έχουμε ακόμα μία παρέμβαση, δεν είναι το τέλος ε, της ε, ακρόασης. Ε, μήπως η κυρία Μέροφ μπορεί να απαντήσει. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Έχω σημειώσει ορισμένα πράγματα που χρήζουν διευκρινήσεως μετά από τις ερωτήσεις σας. Ένας εκ των ευρωβουλευτών αναφέρθηκε στο γεγονό ότι ορισμένοι έχουν δυσκολία να κοιμηθούν μια εβδομάδα μετά από την αλλαγή της ώρας. Εμείς το έχουμε μελετήσει με καμιά πενηνταριά ανθρώπους. Κάποιοι που έχουν ενωρίς χρονότυπο, ας το πω έτσι, έχουν λιγότερες δυσκολίες και προσαρμόζονται σχετικά εύκολα και γρήγορα με τη νέα ώρα κάποιοι που έχουν διαφορετικό χρονότυπο, πιο αργό, πιο, πιο, ε, κοιμούνται πιο αργά, πούμε. Αντιμετωπίζουν τις σχέδιες για πολλές εβδομάδες μετά από την αλλαγή της ώρας. Είναι λοιπόν πιο επίμονο από την εντύπωση, από αυτό που έχουμε την εντύπωση ότι είναι. Αναρωτηθήκατε εάν προτείνω να παραμείνουμε στην χειμερινή ώρα. Ναι, αυτό προτείνω στην βάση συμπερασμάτων της χρονοβιολογικής έρευνας. Σε αυτό διηλίζω ολόκληρη όλα τα συμπεράσματα της έρευνας. Ο συνάδελφος από εδώ διερωτήθηκε γιατί δεν έχουμε ακούσει περισσότερα για αυτά τα πράγματα νωρίτερα. Η χρονοβιολογία τώρα αρχίζει να απογειώνεται ως επιστήμη και ολόκληρος ο τομέας των επιστημών της ζωής δεν είχε ιδέα πόσο σημαντικό είναι το βιολογικό ρολόι. Το βιολογικό ρολόι μετρά όλες αυτές τις λειτουργίες του σώματός μας και τις προσαρμόζει σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Διότι η εξέλιξη έχει καταλήξει ότι αυτή είναι η καλύτερη, η ιδανική στιγμή για να λάβει η χώρα τη συγκεκριμένη λειτουργία. Όταν τα ανατρέπουμε αυτά τα πράγματα, μπορούμε βέβαια να συνεχίσουμε να λειτουργούμε. Αισθανόμαστε ίσω και καλά, ίσω λίγο κουρασμένοι, ίσω να μην μπορούμε να απαντήσουμε πολύ γρήγορα σε ερωτήσει. Κάποιε μικρέ αλλαγέ ίσω σημειώνονται, αλλά είναι μικρέ αλλαγέ που φαίνεται για παράδειγμα στη βάση της επιδημιολογικής μελέτης για το κοινωνικό jet lag, όλες αυτές οι μικρές αλλαγές έχουν ωστόσο σωρευτικό χαρακτήρα. Φτάνει αυτό το κοινωνικό jet lag να είναι μια νόσος των μικρών επιδράσεων. Υπάρχουν και οι νόσοι των σοβαρών επιδράσεων. Αν έχετε για παράδειγμα μία μεταλλαγή του ε, γονιδίου του Χάντιγκτον θα καταλήξετε να έχετε την νόσο του Χάντιγκτον. Εδώ όμως πρόκειται για πολύ μικρές αλλαγές, μικροί εντός εισαγών τραυματισμοί για πολύ μεγάλο διάστημα που ενδέχεται στο τέλος να οδηγήσουν σε νόσο. Αυτού του είδους νόσος είναι αυτό το κοινωνικό jet lag και εμφανίζεται με διάφορους τρόπους. Καρδιακές παθήσεις, παθήσεις του μεταβολισμού, του ανοσιολογικού, κάποιοι καρκίνοι. Διότι το σιρκαδιανό αυτό ρολόι ε, ορίζει όλες αυτές τις λειτουργίες. Αυτά σας δίνω τώρα ως ιστορικό. Έχω συντάξει λευκή βίβλο που εμείς οι χρονοβιολόγοι έχουμε λοιπόν συντάξει ένα έγγραφο για λογαριασμό σας. Θα βάλουμε τον σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της σημερινής συνεδρίασης είναι μια σελίδα όπου περιλαμβάνει με μεστό τρόπο όλα αυτά τα συμπεράσματα των μελετών μας ως χρονοβιολόγων. Πόσοι τώρα επηρεάζονται ή πόσοι θίγονται ή πόσοι πλήττονται καλύτερα. Όσοι αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν ξύπνητήρι πάσχουν από κοινωνικό jetlag. Άρα 80%. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι μεταξύ των ε, νεαρών, των εφήβων. Τώρα ποιο είναι το ιστορικό της εισαγωγής της θερινής ώρας. Δεν μπορώ να σας μιλήσω με καμιά αυθεντία. Έχω διαβάσει όμως κάποιες ιστορικές αναφορές και μια ιστορία που άκουσα ήταν ότι ήταν ένας Βρετανός αρχιτέκτονας ο οποίος πήγαινε στο Λονδίνο καθημερινά και διαπίστωσε ότι το πρωί που πήγαινε με το τρένο στο Λονδίνο είδε ότι οι κουρτίνες των σπιτιών ήταν κλειστές για να μπορεί ο κόσμος να κοιμάται επειδή είχε φως έξω. Θεώρησε λοιπόν ότι αυτό είναι μια περιττή σπατάλη ηλιακού φωτός. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Αλλά βέβαια δεν είναι επιστημονική θεμελίωση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Η άποψή μου για την νομική βάση ε, αφορά δύο σημεία εάν ε, όντως ε, είναι σημαντικό να κερδίσουμε αυτό το πρωινό φως και εάν και κατά πόσον ε, το, η, η ενιαία αγορά μπορεί να κερδίσει κάτι από αυτό το Save Daylight. επί του δεύτερου στοιχείου έχουμε την πρόσφατη νομολογία του δικαστηρίου και ακριβώς εκεί είπα ότι η οδηγία δεν είναι πιστική όσον αφορά την αιτιολόγησή της. Πολλά είναι τα στοιχεία τα οποία αφορούν το Daylight Saving Time ε, και δεν είναι σαφής ε, η επιλογή της νομικής ε, βάσης όσον αφορά αυτήν την εναρμονισμένη καταγραφή της της θερινής ώρας και ενδεχομένως αντί για εναρμόνιση μπορεί να αποτελεί και ένα στοιχείο αθέμη, της τρέβλωσης της εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τα θέματα λοιπόν του δεύτερου γύρου. Τέλος. Αλλά όχι έσχατος. Ο δόκτωρ Βούντερλιχ της Γερμανικής Ένωσης Βιομηχανιών Ενέργειας και Ήδατος από το Βερολίνο. Δέκα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, πρώτα σας ευχαριστώ πολύ που μου επιτρέπετε να συμμετάσχω στην ακρόαση από πλευράς του κλάδου ενέργειας. Λέγομαι Βούντερλιχ, Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Ένωσης ε, Ενέργειας και Νερού και εκπρόσωπος εδώ στις Βρυξέλλες. Θέλουμε να ρίξουμε λίγο φως στο θέμα από την άποψη της ενέργειας. Η τα διαθέσιμα δεδομένα δεν είναι ούτε εκτεταμένα, ούτε και πλήρως ικανοποιητικά, ούτε καν επίκαιρα. Σε ό,τι αφορά την τεχνολογική καινοτομία της παραγωγής ενέργειας έχουν προκύψει νέα πλαίσια που θα πρέπει να μελετηθούν τουλάχιστον εμπειρικά, αλλά θα επανέλθω σε αυτό. Η θερινή ώρα υπάρχει από το 1980 στη Γερμανία τότε κάτω από την επίρρεια της ενεργειακής κρίσης το, της δεκαετίας του 70 για να εξοικονομηθεί ηλιακό φως. Το 1996 γίνεται προσπάθεια στη βάση οδηγίας ευρωπαϊκής ρύθμισης, νομίζω στη βάση μιας μελέτης που συμμετέσχουν εμπειρογνώμονες ενδιαφερόμενοι και χωρισμένοι. Με την εισαγωγή της θερινής ώρας αναζητήθηκε, ή μάλλον επιζητήθηκε η επιζητηθηκε η λειτουργία της ενίας αγοράς, ιδίως στον τουρισμό, στην ε, γεωρική οικονομία και στις μεταφορές. Δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η θερινή ώρα ε, διευκολύνει κάποιους να βγαίνουν το βράδυ, αλλά Δεν υπάρχουν μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις θερινής ώρας στο περιβάλλον. Η θερινή ώρα επέτρεψε κάποιες εξοικονομήσεις ενέργειας, διότι αφού υπάρχει περισσότερο φως το βράδυ δεν ανάβουν τόσο νωρίς τα φώτα. Αυτές όμως οι εξοικονομήσεις εξισορροπούνται από το ότι η θέρμανση αρχίζει να λειτουργεί το πρωί νωρίτερα. Και βέβαια υπάρχει και περισσότερη κυκλοφορία αυτοκινήτων το βράδυ. Επομένως, οι εξοικονομήσει αυτές ούτω ή άλλως είναι δύσκολο να υπολογιστούν και εν πάση περιπτώσει είναι περιορισμένε. Οι επιπτώσεις λοιπόν της θερινής ώρας είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Από την άποψη τώρα της ενέργειας η θερινή ώρα αμφισβητείται. Ποτέ δεν μπόρεσε να αποδειχθεί κάποια σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας το αρμόδιο Ομοσπονδιακό Υπουργείο γίνεται κάποια εξοικονόμηση στο ηλεκτρικό ρεύμα το βράδυ, από την άλλη μεριά όμως, όπως είπα, λειτουργούν οι θερμάνσεις νωρίτερα το πρωί. Υπάρχει και έρευνα του Πολυτεχνείου του Μονάχου του 1983, μικρο και μακροοικονομική ανάλυση της θερινής ώρας στην οικονομική ζωή. Εκεί λένε ότι είναι τόσο μικρή η επίδραση αυτή που είναι αμεληταία. Και από το 1994 παρόμοια μελέτη της προκατόχου μας ενώσεως ε, δεν έχει διαπιστώσει σημαντικές εξοικονομήσεις. Το 2007 κατέθεσε ανακοίνωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσίευσε ανακοίνωση δηλαδή, με πιο σύγχρονα δεδομένα. Εγώ θα πάρω μόνο ένα παράδειγμα. Στην Βουλγαρία διαπιστώθηκε για παράδειγμα ότι η εξοικονόμηση είναι της τάξης του 0,01% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην ε, ε, χώρα. Στη Γαλλία ήταν το 0,014%. Εξοικονομήθηκε λοιπόν κάποιο ηλεκτρικό ρεύμα. Βεβαίως δεν ήταν εκεί οι τεχνικές δυνατότητες όπως είναι σήμερα ήταν λοιπόν πολύ μικρές οι επιπτώσεις. Και στην Εσθονία έχει γίνει μια σχετική μελέτη, όπου το 2000 και 2001 η κατανάλωση των ε, νοικοκυριών ήταν διαφορετική το καλοκαίρι από το χειμώνα. Προφανές. Δεν υπάρχει εν τέλει μεγάλη διαφορά. Πέραν τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Υπάρχει όπως φαίνεται μελέτη από τις ΗΠΑ η οποία θεωρεί μάλιστα καταλήγει ότι υπάρχει μάλιστα αρνητική επίπτωση στην εξοικονόμηση από την πολιτεία Ινδιάνα και από με, μελέτη έρευνα μάλλον σε 7 εκατομμύρια νοικοκυριά είδαν ότι με τη θερινή ώρα αυξάνεται η κατανάλωση κατά 4% πιθανότατα λόγω της θέρμανσης καθώς επίσης και της λειτουργίας των ε, μηχανημάτων κλιματισμού τα ζεστά βράδια. Και από την Αυστρία για το 2013 έρευνα που δείχνει παρόμοια πράγματα. Λέει η ε, αυστριακή έρευνα ότι πιθανώς θα υπάρξει ένα όφελος της τάξης των 4 εκατομμύριων ευρώ τον χρόνο διαρκώς στη θερινή ώρα. Τώρα βέβαια σε ποια βάση έχει γίνει αυτός ο υπολογισμός δεν εξηγείται. Τώρα αυτό που οφείλει να διαπιστωθεί είναι ότι η αλλαγή της ώρας σε ό,τι αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας δεν έχει προσφέρει καμία ωφέλεια. Κάποια εξοικονόμηση υπάρχει αλλά όπως είπα αυτή εξισορροπείται αρνητικά από την ε, νωρίτερη λειτουργία των θερμάνσεων. Ήδη εμείς ως Ένωση έχουμε υποβάλει και σχετική έκθεση από το 2004 βρήκαμε ότι η εξοικονόμηση στα γερμανικά νοικοκυριά ήταν της τάξης του 8% πιθανόν θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη εξοικονόμηση με την χρήση σύγχρονων ε, λαμπτήρων καθώς και ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Τώρα επανεξετάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οδηγία για τη θερινή ώρα. Θα πρέπει να γίνει αυτό στην βάση επίκαιρων επιστημονικών ερευνών. Όχι μόνο για την εξοικονόμηση της ενέργειας, να ληφθεί υπόψη η επίπτωση και στην τροποποιούμενη παραγωγή της ενέργειας, διότι υπάρχει και η ενέργεια, η παράγεται από φωτοβολταϊκά τόξα. Πρέπει να δουν και ποια θα είναι η ωφέλεια από την χρήση της ε, ενέργειας αυτής. Μπορεί λοιπόν η ηλιακή ενέργεια να ενσωματωθεί στο σύστημα της παραγωγής ενέργειας. Εδώ χρειάζεται ακόμα πολύ έρευνα. Θα ήθελα ολοκληρώνοντας να σας παρακαλέσω να εξετάσετε ότι οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να ληφθεί στην βάση επιστημονικών ερευνών, διότι όπως είπα η μέχρι τώρα ρύθμιση δεν έχει αποφέρει ουσιαστικά καμία βελτίωση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ αγαπητή κυρία. Τώρα έχει έρθει η ώρα για να υποβάλλετε ερωτήσεις στον τελευταίο μιλητή. Εσείς κύριε Ρόιλ. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που έχουν σημασία. τονίσατε την αρχή, ότι η αρχή όλης αυτής της υπόθεσης ήταν ότι σε περιόδους πετρελαϊκής κρίσης πρέπει να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Αυτό το καταλαβαίνω. Εάν πάντως μετά από σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και σήμερα πάλι φαίνεται ότι δεν συμβαίνει τελικά αυτή η εξοικονόμηση ενέργειας και ευχαριστώ που τονίσατε ότι υπάρχουν άλλες τεχνικές δυνατότητες για την εξοικονόμηση της ενέργειας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος δύο φορές το χρόνο να κάνουμε αυτή την αλλαγή. Μιλήσατε και για αυτή την δημοσκόπηση που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2007 διότι η ψήφιση οδηγίας απαιτεί και διαβούλευση που δεν προσπάθησαν να την αποφύγουν τότε. Έγινε όμως. Και εσείς είπατε και ορισμένα παραδείγματα από αυτήν. Νομίζω όμως ότι ήταν όντως ευρύτατη και ήδη σε καμία χώρα τότε δεν μπορούσε να μετρηθεί η αδίποτε εξοικονόμηση. Μόνο που, όπως φαίνεται, καμιά χώρα μέλος και ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν καμιά διάθεση να ξεκινήσουν μια τροποποίηση του καθεστώτος τότε. Γι' αυτό ρωτώ. Βασιστήκατε κυρίως σε γερμανικά νούμερα, διότι βεβαίως γι' αυτά είστε αρμόδιος. Τα νούμερα του 2007 που έχει υπόψη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνουν ωστόσο ότι τα νούμερα αυτά που ισχύουν για τη Γερμανία είναι παρόμοια και σε άλλες χώρες μέλη. Κάνατε και μια σύγκριση με την Αμερική που είναι διαφορετική η κατάσταση αλλά πάντως και εκεί η κατάσταση έρει την ισχύ του επιχειρήματος εξοικονόμησης. Λίγο πολύ επομένως έχει ήδη αποδειχθεί ότι είναι τελώς άσκοπη η αλλαγή της ώρας. Εσείς κύριε Νίμπλερ. Ευχαριστώ και εγώ επιθυμώ να ευχαριστήσω τον δόκτωρα Βούντερλιχ για τις ε, εξηγήσεις του. Συμφωνώ απόλυτα στην ουσία με τα όσα είπε ο κύριος Ρόιλ, ότι δηλαδή το πλεονέκτημα ή τέλος πάντων η αιτιολογία για την οποία ψηφίστηκε το 2007 η οδηγία να εξοικονομηθεί δηλαδή ενέργεια προφανώς δεν προέκυψε αυτή η ωφέλεια άρα δεν βλέπω καμία, κανένα νόημα να εμένουμε στην οδηγία αυτή ανεξάρτητα και από τις αρνητικές επιπτώσεις που εξήγησαν άλλοι παρεμβάντες πριν σε ό,τι αφορά τον βιορυθμό, το βιολογικό ρολόι του καθενός και ούτω Επομένως, τώρα δεν έχω άλλε ερωτήσει, αλλά αυτό που με απασχολεί ακόμη είναι, και δεν ξέρω ποιο μπορεί να μα το διευκρινίσει αυτό, είναι τι κοστίζει η αλλαγή της ώρας στην Ευρώπη. Εκτός από τις επιπτώσεις που έχει, τι, τι κόστος έχει αυτή η αλλαγή των ε, δρομολογίων, των τρένων, των ε, ωραρίων λειτουργίας κτλ. Η παράκλησή μου προς εσάς κύριε Πρόεδρε, μετά την σημερινή ακρόαση να δοθεί μια συνέχεια. Ποια θα είναι η μορφή της συνέχειας αυτής, να το σκεφτείτε εσείς, ίσως και να συζητήσετε και με τους συντονιστές, γιατί έχουμε και την μονάδα αξιολόγησης, ας ανατεθεί σε αυτήν. Δεν ξέρω ποια συνέχεια θα πρέπει να δοθεί, δηλαδή αν θα γίνει επερώτηση, αν θα αναλυθεί κάποια έκθεση πρωτοβουλίας. Όμως έδειξε η σημερινή συζήτηση Δεν άκουσα και κανέναν να συνηγορήσει υπέρ της αλλαγής της ώρας. Όλοι οι συνάδελφοι είπαν ότι υπάρχει ανάγκη να αναλυφθεί δράση. Γι' αυτό και παρακαλώ να προωθήσετε και άλλες πρωτοβουλίες ώστε να μην αρχιοθετηθεί το θέμα, αλλά να προχωρήσει. Εσείς κύριε Βούντερη θέλετε να απαντήσετε. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα γερμανικά όμως αφού άλλωστε με ρωτήσατε στην ε, γερμανική γλώσσα. Όποιος εξετάσει την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την έννοια της οικονομίας της ενέργειας είναι σαφώς απαραίτητο να υπάρχει ενιαία ρύθμιση. Δεν μπορώ να θεωρήσω ότι έχουν προκύψει εξοικονομήσεις ενέργειας. Τώρα, εν ώψη των τεχνολογικών εξελίξεων νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια συστηματική έρευνα που δεν έχει γίνει ποτέ ως τώρα. Σήμερα υπάρχουν σημαντικότατες τεχνολογικές εξελίξεις στην αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας, στα φωτοβολταϊκά κτλ. Είπα ότι έχω ορισμένα νούμερα για τη Γερμανία. Έχω κάποια νούμερα από την ισχνή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι να τροποποιηθεί η οδηγία, αλλά από την άποψη της εξοικονόμησης της ενέργειας, και αυτό είναι το δικό μου χωράφι, δεν έχει αποδειχθεί ότι έχουν προκύψει οποιασδήποτε της ενέργειας, αυτό το επιβεβαιώνω. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Πριν ε, ολοκληρώσουμε αυτήν την ε, ακρόαση, θα ήθελα να πω ότι είναι εδώ μαζί μας ε, ο κύριος Σίλερ, γερουσιαστής ε, στη Δημοκρατία της Τσεχίας, ο οποίος θα ήθελε, είναι συντάκτης της έκθεσης για μία ενιαία ώρα και θα ήθελε να μας πει ορισμένα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου λύγετε το λόγο και ε, που μου δίνετε και την ευκαιρία να παρίσταμε στην ακρόασή σας. Να ευχαριστήσω την κυρία Σόιντροβα και τον Παύλ Σφόμποντα, οι οποίοι με βοήθησαν πάρα πολύ ε, κατά την επίσκεψή μου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εγώ ασχολούμαι με το θέμα αυτό εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και έχω μερικά σχόλια. Το θέμα ετέθη πέρσι όταν ε, αιώνα, ε, όταν ε, ο Φραγκλίνος εισήγαγε την ώρα, την θερινή ώρα, ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, ο Χίτλερ έκανε το ίδιο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για να έχει τη δυνατότητα ε, οι μάχες να κρατάνε περισσότερο. Η θερινή ώρα εισήχθη τη δεκαετία του 70 στην κομμουνιστική Τσεχία για να ε, Τσεχοσλοβακία για να ε, υπάρχει περισσότερο φως όμως αυτό είναι αντίθετο με την ανθρώπινη, αυτό είναι η ανθρώπινη φύση ουσιαστικά, η οποία μερικές φορές νομίζει ότι είναι ισχυρότερη από την ίδια τη φύση και ότι μπορεί να παίρνει αποφάσεις αντί αυτής. Η καθηγήτρια Ινέροβα στην τσεχική ε, δημοκρατία έχει καταλήξει στα ίδια συμπεράσματα με αυτά της καθηγήτριας ε, Μέρο και εγώ πολλές φορές ε, αναφέρομαι στα πορίσματα αυτά δεδομένου ότι κανένας δεν κερδίζει τίποτα και 20% του πληθυσμού ε, αναστατώνεται από την αλλαγή της ώρας. Νομίζω ότι το συντομότερο, ε, όσο το συντομότερο την καταργήσουμε αυτή την αλλαγή της ώρας, τόσο το καλύτερο. Όσοι πάσχουν από σύνδρομο Down υποφέρουν ιδιαίτερα και μάλιστα για μεγαλύτερο χρονικό ε, διάστημα. Έχουμε φίλους, συναδέλφους που πάσχουν από σύνδρομο Down και υποφέρουν ιδιαίτερα αν μας ε, απασχολεί αυτό, αν ενδιαφερόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε κάτι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβει δράση. Εμείς θα συνεχίσουμε την εκστρατεία μας στην τσεχική δημοκρατία και θα προσπαθήσουμε να πείσουμε την κυβέρνηση να ε, καταργήσει την αλλαγή από τη χειμερινή στη θερινή ώρα. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο. Να επισημάνω ότι ο Βενιαμίν Φραγκλίνος ήταν περίφημος ως early chronotype. Ήταν, ε, ο χρονότυπος του ήταν δηλαδή ε, νωρίς. Ζητώ συγγνώμη γιατί είναι και συμπατριώτης μου. Okay. Uh, I think... Uh, Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος. Πιστεύω ότι τώρα έφτασε η ώρα να ευχαριστήσω τους έγκριτους ε, ε, ομιλητές μας ε, που μπήκαν στον κόπο να έρθουν και να μας ενημερώσουν. Σας ευχαριστώ επίσης, ευχαριστώ τους συναδέλφους γιατί με στήριξαν ε, στην οργάνωση αυτή της κοινή ακρόασης. Όταν ε, πρώτα έριξα την ιδέα δεν ήταν ε, όλοι έτσι πολύ θετικά διακείμενοι απέναντι στην ιδέα αυτή για να το πω διπλωματικά. Όμως νομίζω ότι πολλά μάθαμε από τους ομιλητές μας σήμερα και το βέβαιο είναι ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να μελετούμε το νομοθέτημα αυτό. Θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε ναι, συζητήσαμε μάλιστα ε, σήμερα το πρωί στους συντονιστές της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων και ε, συμπεράναμε για την ώρα ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μία προφορική ερώτηση προς την Κομισιόν στην επόμενη Ολομέλεια. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει έναν τρόπο επιτάχυνσης, ας πούμε, ε, της διαδικασίας. Φυσικά η κυρία Νίμπλερ έχει δίκιο όταν λέει ότι ε, μια άλλη επιλογή για το μέλλον θα μπορούσε να είναι η, η έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.